Good morning, everybody. I will start uh, our meeting, which... Uh, Καλημέρα σε όλους. ξεκινάει η συνεδρίασή μας η οποία θα κρατήσει σήμερα και αύριο. Λοιπόν, να σας δώσω καψιλοφορίες πρώτα. Σημείο 8. Προστασία του ευρώ. Με συγκεκριτή την κυρία Μακιντάιρ έχει αναβληθεί. Επίσης, και η, ψήφος, ε, η ψηφοφορία επί του σχεδίου ψηφίσματος για τις εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης Ρωμά έχει αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση στις 5 Δεκεμβρίου. Αυτές είναι οι αλλαγές ε, στην ημερήσια διάταξη. Αν συμφωνείτε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ναι, για τη γλώσσα τώρα. Σήμερα δεν έχουμε φιλανδικά και ουγγρικά. ευτυχώς Και σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Αν συμφωνείτε εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Της 29ης και 30ης Μαΐου, της 6ης Ιουνίου, 19ης και 20ης Ιουνίου, 20 ης Ιουνίου, 16 και μέχρι 18 ε, Σεπτεμβρίου. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι αύριο στη λέξη της συνεδρίασης τα πρακτικά εγκρίνονται. Τώρα, το τι γίνεται με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. ή ενδοετερικές μεταθέσεις. Είχαμε χτες ε, έναν διάλογο, θα δώσω όμως το λόγο στον κύριο Γιακολίνη να μας ενημερώσει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χθες ε, στο Συμβούλιο είχαμε τριμερή διάλογο για το θέμα αυτό για το ICT και είχαμε προδιορίσει και το άλλο το θέμα για τους εποχιακά εργαζόμενους και το Συμβούλιο μαζί με μας προσπαθεί να καταβάλει μια κοινή προσπάθεια για να συμφωνήσουν τα θεσμικά όργανα και αυτό όσο γίνεται συντομότερα. Και χθε ήταν που έγινε κάτι το θετικό για μας. Πρώτα απ' όλα να δούμε πώς ε, οι εθνικές ε, μέθοδοι δεν θα ισχύουν πια και η διαδικασία από τη στιγμή που θα ιωτηθεί θα πρέπει να αφορά όλα τα κράτη-μέλη για ένα μέτρο ομοιόμορφο κοινό. Και από τη μία εταιρεία στην άλλη μεταφορά ε, έχουμε μια μείωση χρονική, μόνο έξι μήνες ε, και κοιτάζουμε να δούμε και τα όργανα πώς θα αντιδρούν για να μπορούν να δίνουν μια άδεια μαζί και με, τους, ε, με τα μέλη της οικογένειας και να μπορεί να εξεταστεί καλύτερα ένα φάκελος που χρειάζεται από τους ειδικού μια γνώση και να μπορούν ε, να έχουν μαζί και τα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτά σχετικά με την κινητικότητα ατόμων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στη αρχιπρόθεσμη και στη μακροπρόθεσμη. Μερικά σημεία όμως θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε με το Συμβούλιο. Και σαν Κοινοβούλιο είπαμε όχι ε, ότι υπάρχει μια οικονομική ευθύνη για την ανάλυση των εξόδων αυτών και εμείς θέλουμε κάτι το καλύτερο, πιο εύκαμπτο και αποτελεσματικό. Μερικά θέματα ακόμα για τις ποσοστώσεις και για την προσβασία, όχι αυτά που προβλέπονται από την Λισαβόνα, αλλά με διάφορες άτρες δυνατότητες στις οποίες διαφωνούμε και τα ζητάει όμως το Συμβούλιο. Υπήρξε μια έντονη διαπραγμάτευση Σίγουρα όμως ήταν κάτι το θετικό και με τους κοιόδης συγητές που πήραν το λόγο, Μόλντερ και Σερζεντίνη και με τη γραμματεία, τη βοήθειά της. Για το άρθρο 14 έχουμε ένα θέμα ακόμα, για άλλα θέματα, για αρμοδιότητες της ε, Επιτροπής Σέμπολ. και χθες το βράδυ ε, στο Γιακουρσάρι που η Επιτροπή της είναι αρμόδια για αυτά, για την Επιτροπή και να μπορέσει να προωθήσει όσο γίνεται ταχύτερα μια συμβαστική λύση, να υπάρξει δυνατότητα το θέμα αυτό να κλείσει η έκθεση αυτή μέσα σε αυτό το εξάμεινο Λιθουανικής Προεδρίας ή τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Ελληνικής Προεδρίας στη συνέχεια ώστε να υπάρξει μια σχετική έγκριση το Φεβρουάριο και Μάρτιο και να μπορούμε έτσι να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα σημαντικό εργαλείο στην Ευρώπη που να συμφιλειώσει όχι καλύτερα την αγορά εργασίας με την αναζήτηση εργασίας από άτομα από τρίτες χώρες αλλά με αρισμένα ειδικά προσόντα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αφού ψηφίσαμε χτες ε, για τα θέματα που αφορούσαν δικαιοσύνη και σήμερα για τον Περικλή 2020 οι φάκελοι σχετικοί θα πάνε στο τελικό γύρο διαπραγματεύσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε βεβαίω συνομιλίες για τους τρεις συγκεκριμένους κανονισμούς, δηλαδή τα σύνορα, την αστυνομία και το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και μετά θα συζητήσουμε το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης την επόμενη εβδομάδα και τον οριζόντιο κανονισμό. Το ζήτημα λοιπόν των πράξεων κατεξιοδότηση ήταν στην ημερήσια διάταξη υπό την Προεδρία της Επιτροπής μας, του κυρίου δηλαδή Λόπεζ Αγγιλάρ, ο οποίος ε, έχει την πεποίθηση πως οι συγητές θα διαπραγματευτούν για αποτελέσματα τα οποία θα εφηρεμίζονται με αυτά τα οποία ζήτησαν οι πρόεδροι στη διάσκεψη των πρόεδρων. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ελπίζουμε να γίνει την ίδια μέρα δηλαδή πριν από το τέλος του χρόνου. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, η Συγητής είναι ο κύριος Μέλο, ο οποίος όμως δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έρθει στις 10 η ώρα από ό,τι μου είπαν. Οπότε διακόπτουμε για λίγα λεπτά. Μέχρι να έρθει ο εισηγητής. Ελπίζω να έρθει στην ώρα του. Take your seat, Mr. Καθίστε. Τελείωσαν οι συνάδελφοι το διάβασμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Κύριε Μέλλο, είμαστε στο σημείο 5. Εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την γνωμοδότησή σας για την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Αλλά μου είπαν ότι χτες ο ε, τριμερής διάλογος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας ε, ολοκληρώθηκε και εσείς θα θέλετε να πείτε λίγα λόγια ως συγητής. Μια ναι, λοιπόν που ήταν αυτό στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ενημερώστε μας πρώτα και μετά θα περάσουμε στη γνωμοδότηση. ήθελα να πω το εξής. Ναι, πραγματικά χθες ε, πετύχαμε μία συμφωνία στον τριμερή διάλογο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ήταν πολύ σημαντική έκθεση και έτσι σε αυτό το κοινό χώρο με μια ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, κεφαλαίων, υπηρεσιών κλπ μπορούμε να έχουμε και ένα κοινό χώρο για τη δικαιοσύνη. Με μια εγγύηση ότι τα μέσα αυτά έρευνας για την εγκληματικότητα να αποτελούν μέρη μιας αμοιβαία αναγνώρισης και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις διάφορες χώρες σε σχέση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Είναι λεπτά θέματα και είχαμε έντονες διαπραγματεύσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις και τελικά είχαμε την έγκριση αυτή στα πλαίσια του ε, τριμερής διαλόγου. Αυτή είναι η ενημέρωση που ε, θα ήθελα να σας κάνω. Ευχαριστώ. Και τώρα μπορείτε να περάσετε στη σχέδιο νομοδότησης που προετοιμάζει η ΛΥΜΠΕ για την ΑΦΚΟ σε σχέση με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Ακούστε, το ε, χρησιμότερο που θα μπορούσα να σας πω είναι κάπως μικρό σε σχέση τουλάχιστον με αυτά τα οποία συντάχθηκαν καλύτερα να μπορούσα να σας μιλήσω το τι θεωρώ ότι θα μπορούσα να παρουσιάσω στην ΑΦΚΟ που είναι και αρμόδια επί της ουσίας και να ενταχθεί στο κείμενο ψηφίσματος που εγκρίθηκε μόλις. Έχουμε πέντε βασικά σημεία. Να πενθυμίσουμε για το νομοθετικό πλαίσιο, εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι ενισχύει τις ρυθμιστικές του αρμοδιότητες και θα ήθελα να τονίσω ότι τα νομοθετικά ε, μέτρα ε, εγκρίνονται με μέσω μιας κανονικής τακτικής νομοθετικής διαδικασίας και να δούμε τώρα και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στη συμπερίληψη στον χάρτη της Λισαβόνας. Τι σημαίνει αυτό είναι κάτι δεσμευτικό νομοθετικά και ο χάρτης αυτός θα πρέπει να γίνεται σεβαστός από τη στιγμή που εφαρμόζει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύο θετικές πτυχές που θα ήθελα να τονίσω για την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Ταυτόχρονα όμως και άλλα σημεία που θα πρέπει να παρατηρήσουμε πιο συγκεκριμένα για να δούμε τρία σημεία. Να σας υπενθυμίσω, υπενθύμισα ήδη, ότι μέσω της συνθήκης η Επιτροπή έχει κατεξοδότηση ε, εξουσίες ε, και η Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στις πράξεις ε, εκτέλεσης και της κατεξιοδότησης. Και αυτό, όπως αναφέρονται, πέρα από αυτά που αναφέρονται στις συνθήκες, θα πρέπει η Επιτροπή να ε, ενημερώνει τακτικά για τις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις διεθνείς συμφωνίες όταν έχουν να κάνουν και με θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Και δυστυχώς σημειώνεται έλλειμμα παρά την συνθήκη της Λισαβόνας δεν σημειώθηκαν βελτιώσεις και κάτι συμπέρασμα. Θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο σε ορισμένε περιπτώσει να έχει ανοιχτέ συνεδριάσει όπω ομάδε εργασίε, Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων κλπ. για να μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό σημαίνει και με τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Υπάρχει μια συνεργασία έντιμη ξεκαθαρή ανάμεσα στα όργανα που συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή. Αυτά θα ήθελα λοιπόν να τονίσω και από τη στιγμή που συμφωνούν οι συνάδελφοι να δούμε την προθεσμία για τις τροπολογίες 17 Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι είναι κάτι το λογικό σαν προθεσμία. Έτσι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Μέλα. Θα ήθελε μήπως το λόγο κάποιος συνάδελφος. Εάν όχι, τότε, όπως σωστά προτείνατε, στις 17 Δεκεμβρίου θα είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και προχωράμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης, αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης με εισηγητή, εισηγητρία την Βαρόνη Σαρα Λάτφορτ, όπως γνωρίζουμε Η απόφαση πλαίσιο του 2002 είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις και είναι η πιο ουσιώδης εφαρμογή της αρχής της ε, αμοιβαίας αναγνώρισης. Ωστόσο, έχουν ανακύψει σημαντικά ερωτήματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της και τον τρόπο εφαρμογή της και χρήστης της. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία να βελτιώσουμε το τρέχον, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Βαρόνι Λάτφορτ, η οποία θα μας παρουσιάσει την ε, σχέδιο γνωμοδότησής της και τις συγκεκριμένες προτάσεις της. Γνωρίζω, με ενημέρωσαν μάλλον ότι έχει διανεμηθεί σε όλες τις γλώσσες αυτό το ε, σχέδιο γνωμοδότησης. Κυρία Λάτφορτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ξεκινήσαμε κάπως νωρίς και δεν πρόλαβα να ενημερωθώ, είπατε ότι δεν διανεμήθηκε λάθος, νόμιζα ότι είχε διανεμηθεί. ναι, όχι, έχει διανεμηθεί σε όλες τις γλώσσες. Και ανησύχησα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Είμαι ευτυχής που μπορώ να παρουσιάσω την έκθεσή μου, που είναι αποτέλεσμα στενή συνεργασία με τους κύριους εισηγητές και εσάς ανάμεσα σε αυτούς κύριε Κάρλ. Ευελπιστώ λοιπόν ότι και στη συνέχεια της διαδικασίας αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί. Έχουμε λοιπόν εδώ μια έκθεση, όχι ιδιαίτερα μακροχελή, τρεις-τέσσερις σελίδες και ένα, μαζί με ένα παράρτημα και την αιτιολογική έκθεση, στην οποία προσπαθούμε να καταγράψουμε τις σημαντικότερες προκλήσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ξεκινώ την εκθεσή μου αναγνωρίζοντας το σημασία της απόφασης πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, ε, την σημασία αυτής της απόφασης για το, τις συνεργασίες σε ποινικέ υποθέσεις και την ε, μεγάλη ε, συνεισφορά που είχε αυτή η απόφαση έτσι ώστε να βελτιωθεί η ταχύτητα της συνεργασιών και των εκδόσεων κτλ. Ωστόσο, σε τομείς όπως η τρομοκρατία, αναφέρομαι στο κείμενο του, της απόφασης πλαίσιο που έχει δημιουργήσει προβλήματα. Τα προβλήματα κυρίως έχουν προκύψει από την εφαρμογή. Δεν μπαίνω σε αυτά τα ζητήματα γιατί θα αποτελέσουν αντικείμενο ε, εξέταση του 2014. Αναφέρομαι ωστόσο στο ζητήματα της αμοιβαία αναγνώρισης και γενικότερα της εξέλιξης του ενίου χώρου δικαιοσύνης στο πάνω μέρος της ε, δεύτερης σελίδας της έκθεσης ε, καταγράφω έναν κατάλογο 10 ανησυχιών, 10 προβλημάτων τα οποία θα σας παρουσιάσω. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει ε, ρητά, προβλέπεται κάποιος λόγος ε, για να απορρίψει μια χώρα ε, ένα αίτημα έκδοσης εντάλματος, ε, εφαρμογής μάλλον εντάλματος σύλληψης επί τη βάση του κινδύνου παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα δημιουργήσει διαφορετικό τρόπο μεταγραφής στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή σε κάποια κράτη-μέλη θα μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η ρητή δυνατότητα απόρριψης για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτό δεν θα δώσει μια ομοιομορφή εικόνα. Δεύτερον, το θέμα των ένδικων μέσων, το δικαίωμα στα ένδικα μέσα σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι όποιοι κανόνες, αυτό επαφίεται στο εθνικό δίκαιο, το οποίο θα δημιουργήσει διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τρίτο πρόβλημα. Δεν είναι σαφές πώς θα ε, συνδέονται το σύστημα Schengen, το πληροφοριακό σύστημα Schengen, σε περίπτωση που υπάρξει απόρριψη εντάλματος, ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψη. Δεν προβλέπεται κάποια αυτόματη διαδικασία ή έστω ημιαυτόματη αυτόματη διαδικασία, δηλαδή. Σε περίπτωση που αποσυρθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη, θα έπρεπε ε, το σχετική εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα Schengen να διαγράφεται, αλλά αυτό δεν προβλέπεται. Επίση, δεν προβλέπεται τι γίνεται σε περίπτωση που απορριφθεί αυτό το ένταλμα σύλληψη. Για παράδειγμα απορριφθεί από ένα κράτο μέλο, αλλά το... η εγγραφή συνεχίζει να υπάρχει στο πληροφοριακό σύστημα Schengen και έχουν υπάρξει περιπτώσει ε, άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από τέτοιε καταστάσει. Τέταρτο ζήτημα είναι κάτι που είναι γνωστό, η δυσανάλογη χρήση του ευρωπαϊκού αντάλλαγματος σύλληψη για πτέσματα ή για μικρή σημασία δικήματα. το οποίο ουσιαστικά οδηγεί σε παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών και σε αυθαίρετε συλλήψει, αλλά επίση και σε μεγάλα έξοδα για κράτη-μέλη. Μετά, δεν είναι σαφή τι σημαίνει για λόγους άσκησης ποινική δίωξης που είναι στο σημείο 1 της απόφασης πλαίσιο. Λέγεται ότι τα εντάλματα σύλληψης χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσαχθούν ε, άτομα ως ύποπτοι ή ως ε, μάρτυρες και όχι για να ασκηθεί εναντίον τους ε, δίωξη στο στάδιο της προδικασίας. Αυτό όμως είναι καταχρηστική χρήση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Δεν είχε δημιουργηθεί για να χρησιμοποιηθείτε είτε στην ε, διερεύνηση μιας υπόθεσης, αλλά κατά τη διάρκεια της άσκησης της δίωξης. Μετά έχω κάποιες ανησυχίες σε σχέση με το χρήση του όρου Judicial Authority, δικαστική αρχή. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του όρου από τα διάφορα κράτη-μέλη. Και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και πρόσφατα μάλιστα έχουν υπάρξει και ε, νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου της ε, Μεγάλης Βρετανίας σε σχέση με τον ορισμό της δικαστικής αρχής της έννοιας αυτής σε σχέση με την Λιθουανία. Μετά υπάρχει το ζήτημα της μη πρόβλεψης για αποζημίωση σε περίπτωση που ε, υπάρξει δικαστικό λάθος. Γνωρίζω περιπτώσεις όπου συνελήφθη λάθος άτομο και κανένα από τα δύο εμπλεκόμενα κράτη-μέλη, ούτε εκείνο που είχε εκδώσει το ένταλμα, ούτε εκείνο που το εκτέλεσε, δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει την ευθύνη και να αποζημιώσει τον παθόντα, αυτόν που ταλαιπωρήθηκε από αυτή τη διαδικασία. Μετά υπάρχει το ζήτημα της υπερβολικά παρατεταμένης ε, προφυλάκησης η προφυλάκηση θα έπρεπε να είναι το τελευταίο, η τελευταία επιλογή, αλλά πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως η πρώτη επιλογή. Ακριβώ επειδή δεν υπάρχει ε, ομοιομορφία. Και επίσης συνδεδεμένο θέμα είναι το ζήτημα των διαφορετικών ε, συστημάτων κράτησης και υποδομών κράτησης στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης, ένα άλλο σημείο που συνδέεται με πολλά από τα προηγούμενα είναι το γεγονό ότι δεν χρησιμοποιούνται επαρκώ τα εργαλεία που ήδη έχουμε στη διάθεσή μα για την αμοιβαία συνεργασία στον τομέα των ποινικών υποθέσεων. Και θα επανέλθω σε αυτό όταν μιλήσω για τι λύσει τι οποίε προτείνω. Στην επόμενη σελίδα, στην πρώτη παράγραφο, υπενθυμίζουμε ότι στην γνωμοδότηση αυτή δεν προσπαθούμε να αναφερθούμε στην ε, λανθασμένη κακή χρήση του Ευρωπαϊκού Αντάλληματος Σύλληψης. Ε, μιας και πρόκειται για ονομοδότηση ιδίας πρωτοβουλίας για νομοθετική πρωτοβουλία, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση του άρθρου 82 να παρουσιάσει μια νομοθετική ε, πρόταση, η σειρά νομοθετικών προτάσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που καταγράφουμε. δηλαδή όλα τα προβλήματα τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την ε, κακή εφαρμογή. Πρώτα απ' όλα, να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα απόρριψη τη εκτέλεση του εντάλματο σύλληψη όταν υφίσταται κίνδυνο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελευταία νέα. Χθε το βράδυ συμφωνήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ε, το, ε, το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Έρευνα και μετά από πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταφέραμε σε αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία, δηλαδή στο ένταλμα έρευνα, να υπάρχει τέτοια ρητή πρόβλεψη. Δηλαδή να δίνεται δυνατότητα στο εκτελών κράτος μέλος να απορρίψει την εκτέλεση του εντάλματο όταν θεωρεί ότι υφίσταται κίνδυνος παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο και να προβλεφθεί κάτι ανάλογο και στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και άλλα παρόμοια στην υπόθεση Ράντα, πριν από ένα χρόνο, μια υπόθεση από τη Ρουμανία, ένα από τα προβλήματα που είχε το εκτελών κράτος μέλος, που δεν είχε τη δυνατότητα να απορρίψει την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, ήταν ακριβώς ότι δεν υπήρχε αυτή η ρητή εφαρμογή, ε, η ρητή αναφορά, συγγνώμη. Θα πρέπει να καλυφθεί λοιπόν αυτό το κενό. Μετά ζητάμε να υπάρχει έλεγχος αναλογικότητας στις αποφάσεις αμοιβαίας αναγνώρισης. Ε, αυτός ο έλεγχος ε, δεν θα πρέπει να γίνεται από το εκτελών κράτος μέλος, γιατί αυτό θα δημιουργούσε μεγάλο βάρος. Θα πρέπει αυτός ο έλεγχος ε, αναλογικότητας να γίνεται από το κράτος μέλος που εκδίδει το ένταλμα. Και να εξετάζονται όλα τα εναλλακτικά μέτρα και επιμένουμε σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης έχει, ε, του έχει δοθεί πολύ μεγάλη βαρύτητα ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία δεν αξιοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Κάτι ακόμα που ζητούμε θα πρέπει να τυποποιηθεί η διαδικασία με την οποία ανταλλάσσουν πληροφορίες τα εκτελούντα και τα, ε, τα ετούν τα κρατη Για, παράδειγμα, το κατά πόσον μια, μια δίωξη είναι έτοιμη να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου. Θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα να ανταλλάσσονται αυτές οι πληροφορίες για να μην γίνεται κατάχρηση του εντάλματος υπερβολικά νωρίς στην όλη ε, δίωξη. θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια τυποποιημένη διαδικασία για να επικυρώνεται από δικαστική αρχή στο ε, κράτος μέλος που εκδίδει το ένταλμα ε, σύλληψης. Υπάρχει επίσης ένα τεχνικό σημείο σε σχέση με ε, τον ορισμό της δικαστικής αρχής. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται τα δικαιώματα άσκησης ενδικών μέσων και ε, αποκατάσταση σε περίπτωση ε, πλάνης. Αυτές είναι οι προτάσεις και οι διορθώσεις που ζητούμε. Ζητούμε να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά της Επιτροπής για όλα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται συστηματική αναθεώρηση, ανασκόπηση των ε, ευρωπαϊκών ανταλμάτων σύλληψης, τα οποία τελικά δεν εκτελέστηκαν και επίσης να προβληφθεί μια διαδικασία για να ε, διαγράφονται αυτά τα στοιχεία, αυτές οι εγγραφές από το σύστημα Schengen και το σύστημα της ε, Ευρωπόλ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων, θα πρέπει να υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση των απορρίψεων. Ε, επίσης όλο αυτό το πλέγμα ε, εργαλείων για την ποινική ε, συνεργασία, είτε πρόκειται για την απόφαση πλαίσιο για την ε, μεταγωγή, την επιτήρηση. Όλα αυτά τα εργαλεία δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε. Και θα πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου το Ευρωπαϊκό Ένταλμα να περιοριστεί μόνο στο σκοπό για τον οποίο προοριζόταν. Αναφέρομαι επίσης στην αποζημίωση σε περίπτωση δικαστικής πλάνης και στη στο σημείο 7 ζητάμε από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο και μεταξύ των εισαγγελέων και των δικαστικών αρχών, αλλά επίσης και των μαχόμενων δικηγόρων, έτσι ώστε να ενημερωθούν καλύτερα για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα αυτό ουσιαστικά ε, βελτιώνει την ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να σπαταλά κανείς χρήματα ε, για να ξεκινά διαδικασία ποινική δίωξη με βάση το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη όταν αυτέ δεν πρόκειται να τελεσφορήσουν. Θα πρέπει να υπάρχει μια εκπαίδευση ε, και των εισαγγελέων και των δικαστών και των δικηγόρων. Γιατί δεν είναι επαρκή η ενημέρωση του κλάδου του δικαστικού για αυτά τα θέματα και ζητούμε επίσης να προβλεφθεί χρηματοδότηση όπως για παράδειγμα σε φορείς όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ποινική Δικαιοσύνη, και προτείνουμε μάλιστα να δημιουργηθεί και ένα ξεχωριστό δίκτυο εκείνων που ασχολούνται με το Ευρωπαϊκό ε, Ένταλμα Σύλληψης, στο οποίο να συμμετέχουν και δικηγόροι. Κάποιοι ζητούν μια διαδικασία πιο θεσμοθετημένη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε κάτι τόσο έτσι ε, περίπλοκο. Ας ξεκινήσουμε με έναν επίσημο δίκτυο. Και τέλος, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα νομικά και οικονομικά εργαλεία που έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η κατάσταση ε, όσον αφορά την προφυλάκηση. Ήταν περιορισμένος ο χώρος που είχα στη διάθεσή μου για την ε, γνωμοδότηση, επομένως δεν μπόρεσα να ε, αναφερθώ όσο αναλυτικά θα ήθελα σε ορισμένα ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά το παράρτημα, ακολούθησα την πεπατημένη όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις ίδιας πρωτοβουλίας και προτείνουμε ορισμένες διατυπώσεις που θα θέλαμε να δούμε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Επιτροπή. Υποδεικνύουμε κάποιες διατυπώσεις. Ε, ευχαριστώ λοιπόν να ακούσω και την άποψη των σκιωδών εισηγητών. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η επόμενη ε, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα σας ε, ζητήσω να είστε αυτό το δυνατόν πιο σύντομοι. Σας πενθυμίζω πως στις 11 η ώρα έχουμε ψηφοφορίες. Ξεκινάμε από τους σκιώδες εισηγητές και μετά θα ακούσουμε τους εκπροσώπους της Προεδρίας και της ε, Κομισιόν. Εγώ είμαι σκιώδες εισηγήτρια για το ΕΛΚ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λάντφορτ για την δουλειά που έκανε. Νομίζω πως είναι πολύ καλό το σχέδιο έκθεσης και βεβαίω αντιμετωπίζει και αναφέρει ξεκαθαρά όλα τα προβληματικά ζητήματα που συζητάμε και που υπάρχουν όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Βεβαίω, συμφωνούμε όλοι πως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο αυτό ένα από τα σημαντικότερα στον τομέα της ποινική συνεργασίας. Οπότε πρέπει να λειτουργεί σωστά και βλέπουμε πως υπάρχουν κενά στην εφαρμογή του. Κενά στην αντίληψη του μέσου αυτό. Συμφωνώ με τον κατάλογο που συνέταξε η συγγήτρια και βλέπω, χαίρομαι που υπάρχει ένα έλεγχος αναλογικότητας, εγώ θα έλεγα μάλιστα διπλός έλεγχος πρέπει να υπάρχει και για τις δύο χώρες και είναι θετικό το ότι περιλαμβάνεται η αποσυρσή του εάν αποσυρθεί για υποχρεωτικούς λόγους. Επίσης σημασία έχει η εκπαίδευση των εθνικών νομικών και δικαστικών, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Και όπως λέει και η παροιμία στη χώρα μου, μην καούν τα χλωρά μας με τα ξερά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ε, βλάψουμε τα εφιστάμενα μέσα. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο θέλει η συγγήτρια για το να βελτιώσει δηλαδή την κατάσταση, αλλά θα τονίσω και τον ρόλο των κρατών μελών και των εθνικών δικαστικών αρχών στην εφαρμογή της ε, οδηγίας πλαισίου και την κύρια δική τους ευθύνη. Αυτά από μένα και το ΕΛΚ Τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Τζίπλ. vielen Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λατφόρτ για την έκθεσή της. Είναι πολύ αναλυτική, νομίζω πως υπήρχε μεγάλη συμφωνία μεταξύ των σχεδόν εισηγητών για το πού βρίσκονται τα προβλήματα στο Ευρωπαϊκό Εντέλμα Σύλληψης. Δεν θα επαναλάβω τα προβλήματα αυτά. Περιγράφονται νομίζω πολύ αναλυτικά. Έχω ένα ζήτημα αρχής εδώ πέρα. Το ένταλμα αυτό υπάρχει από το 2002 και σχεδόν από την αρχή εδώ στο Κοινοβούλιο συζητούσαμε για τα προβλήματα της εφαρμογής. Αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα, εξακολουθούμε να συζητάμε για τα προβλήματα, για τη λανθασμένη χρήση, για το ότι διαρκεί πάρα πολύ η διαδικασία, η χρόνη κράτησης. Τα γράφει τώρα εδώ πέρα το έγγραφο, δεν θα τα ξαναπώ. Το πρόβλημά μου είναι πως αν κάνουμε ό,τι λέει εδώ πέρα δεν θα αλλάξει τίποτα. Συζητάμε εδώ και 10 χρόνια τα προβλήματα στην εφαρμογή. Δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν. Δεν μπορούν. Τι νόημα έχει ένας νέος κανόνας, μια νέα, ένα νέο ένταλμα. Ποιο μεσοπίεση έχουμε για να φροντίσουμε για τη σωστή εφαρμογή. Χθε στην ε, Γιούρη συζητήσαμε το θέμα σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μήπως λοιπόν το πρόβλημα είναι πως τα κράτη-μέλη και άλλα θεσμικά όργανα θέλουν να συντονίσουν ε, καλύτερα τα ζητήματα αυτά, αλλά αντιθέτως δεν ε, δείχνουν τον ίδιο ζήλο για το ε, δικονομικό δίκαιο, για τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Ναι, δηλαδή τα προβλήματα είναι γνωστά, αλλά ποια είναι τελικά η ενδεδειγμένη διαδικασία για να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Για το κουτί της Πανδώρας αναρωτιέμαι τι θα γίνει εάν το ανοίξουμε. Λένε όλοι, υποτίθεται πως είναι ένα καλό μέσο. Ε, τότε θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον όλων να λειτουργεί καλύτερα. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι λίγο περίεργη αυτή η συζήτηση. Δεν έχω καμία λύση αυτή τη στιγμή πως θα μπορέσουμε να το λύσουμε, αλλά... Το σημείο 1 της εισηγήτριας θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε όλοι μαζί. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να μιλήσω Ολλανδικά σήμερα. Είμαι ικανοποιημένη από αυτό το οποίο ανέλαβε να κάνει το Κοινοβούλιο μέσω της κυρίας Λάτφορντ. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να πει το Κοινοβούλιο πως ε, δεν μπορούμε να πούμε πως είμαστε σίγουροι για την μεταχείριση των ε, κατηγορουμένων. Είχα συζητήσει με έναν Ολλανδό, ο οποίος είχε συλληφθεί στην ε, Πολωνία και τελικά κατάφερε μετά από 8 μήνες προφυλάκηση να απελευθερωθεί μόνο αφού έβαλε δικηγόρο και στην Πολωνία και στην Ολλανδία και ήταν υποκράτηση σε πολύ κακές συνθήκες. Οπότε η αναλογικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για να μην μένουν οι άνθρωποι 8 μήνες μακριά από τη χώρα τους, μακριά από την ε, οικογένειά τους και μετά να τους λένε εντάξει όλα καλά τώρα. Επίσης πρέπει να δούμε τις συνθήκες κράτησης έτσι να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε κάθε φυλακή ή κάθε κρατητήριο. Επίσης, πρέπει να δούμε τους ορισμούς του ποινικού δικαίου. Όταν μιλάμε για παράδοση υπόπτων από την Ολλανδία στη Σουηδία για μαλακά ναρκωτικά. Δεν θα περνούσε αυτό το πράγμα από ε, δικαστήριο. Δηλαδή όταν κάτι δεν είναι αξιόπινο στην Ολλανδία αλλά είναι σε άλλη χώρα, τι κάνουμε. Επίσης, η πρόταση που αναμένουμε για την νομική συνδρομή. Πρέπει κάποιος να μπορεί να έχει δικηγόρο και στις δύο πλευρές διαδικασίας. Οπότε στηρίζουμε την πρόταση της κυρίας Λάντφορντ, αλλά θέλουμε να σκεφτούμε περισσότερο τα δικαιώματα των κατηγορουμένων όταν μιλάμε για αυτό το τεστ της αναλογικότητας και θέλουμε επίσης συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία θα φροντίζει οι ύποπτοι να μην ε, πάνε σε ε, προφυλάκηση άδικα και αυτό το τελευταίο έχει μεγάλη σημασία για να λειτουργήσει σωστά. Γιατί ο αλλοδαπός ύποπτο θεωρείται πάντα ύποπτο φυγής. Έτσι. Οπότε δεν τον αφήνουν, αλλά είναι προφυλακισμένος σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κέκοπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε. Να συγχαρώ πρώτα την Βαρόνη Λάντφορντ για τη δουλειά που έκανε. Προφανώς το μέτρο αυτό είναι πολύ σημαντικό και οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα παρά τις ελλείψεις του είναι ένα πολύτιμο μέσο επιβολής του νόμου. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, αποφεύγονται Μακροσκελής ε, διαδικασίες έκδοσης, ειδικά σε περίπτωση διασυνοριακής τρομοκρατίας. Η ταχύτητα είναι μεγάλο προσόν του, ειδικά από όταν ε, ισχύει η ζώνη Σέγγεν, οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, διασυνοριακή εγκληματικότητα, οπότε η έκδοση πήγε από τους 18 μήνες κάποιες εβδομάδες. Και το σημαντικό θέμα εδώ είναι να αναγνωρίσουμε την επιτυχία. Α, ακούγα τους προηγούμενους ομιλητές πως ε, ναι πρέπει να τα έχουμε δει τα ζητήματα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι, ναι, αλλά οπωσδήποτε. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τα στοιχεία. Νομίζω το έχει κάνει αυτό η συγκήτρια. Και να δούμε πού μπορούμε να το βελτιώσουμε. Αυτό το οποίο λοιπόν θα ήθελα εγώ να βελτιωθεί πρώτα απ' όλα είναι το θέμα της αναλογικότητας. Χρειάζεται νομίζω εδώ μεταρρύθμιση. Πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα αναλογικότητας όταν αναθεωρηθεί για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο ορισμός κάποιων αξιόπινων πράξεων εντός του εντάλματος επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες από χώρα σε χώρα. Π.χ. η Η απάτη, παραδείγματο χάρη, μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους. Αυτή τη στιγμή επίση τα δικαστήρια δεν μπορούν να απορρίψουν τα αιτήματα. Αλλά η κρίση της αναλογικότητας είναι στη διακριτική ευχαίρεια βεβαίως του φορέα που θα εκτελέσει το ένταλμα. Δεν υπάρχουν επίσης περιορισμοί στη χρήση και ε, εγγυήσεις και δεν υπάρχει δυνατότητα βέβαιως προσφυγής εναντίον της ε, πράξης αυτής και η της ασφαλείας που λεγόταν δικαστής δεν υπάρχει πλέον. Οπότε κυρία Πρόεδρε, οπωσδήποτε κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Το ερώτημά μου το εξή. Όλοι τα βλέπουμε λίγο πολύ τέτοια πράγματα, σε κάποια άλλα, τα είπε και η συγγήτρια. Εγώ θα ήθελα να είμαι σίγουρος πως θα γίνουν οι αλλαγές που ζητάμε. Ξέρετε, τα παραδείγματα χρήσης ε, του εντάλματος για πτέσματα ε, είναι σαφώς ε, θέμα αναλογικότητας. Πρέπει νομίζω να φροντίσουμε πως τα εντάλματα αυτά δεν θα εκτελούνται όπου υπάρχουν ε, σοβαρές ε, ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, όπως ανέφερε η Σίγητρε και ως νομικός έχω ισχυρή άποψη ε, όσον αφορά την πρόσβαση σε δικηγόρους, πρέπει να υπάρχει πραγματική εκπροσώπηση και στο κράτος ε, έκδοσης του εντάλματος και στο κράτος εκτέλεσης. Οπότε, Συνελώνται η κυρία Πρόεδρε, γιατί βλέπω ότι θα πατήσετε το μικρόφωνο. Στηρίζω την εισηγήτρια και το ένταλμα, αρκεί να γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές και νομίζω πως ε, πρέπει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας να φροντίσει να συνεχίσει να στηρίζει το ένταλμα αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή, αλλά και για τη συνεργασία. Είχαμε, νομίζω, κάποιες αρκετά χρήσιμες συναντήσεις. και είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Έχω κάποιες παρατηρήσεις βεβαίω που θα αναφέρω. Πρώτη, στην πρώτη παράγραφο λέει πως δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή του ιδίου του εντάλματος. Μπορεί βεβαίως κάλλιστα η συζήτηση στο Συμβούλιο να πάει προς την κατεύθυνση που θέλουμε και να υπάρξει ένα τελείως ε, διαφορετικό μέσο. Θεωρώ λοιπόν πως πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ ε, βράχυπρόθεσμων ε, ενεργειών για να αλλάξει το Ευρωπαϊκό Τέλμα Σύλληψη και των λοιπόν που θα είναι μακροπρόθεσμα ή μπορεί να είναι κάποιο διαφορετικό εργαλείο. Μετά κάτω από η μπορει να ειναι καποιο διαφορετικο εργαλειο μετα κατω απο την ρητρα για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε να είμαστε σύμφωνοι με την ΕΣΔΑ, την Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεύτερον, για την αναλογικότητα. Υπάρχει αναλογικότητα βεβαίως και από το κράτος έκδοσης ε, τι γίνεται στην περίπτωση που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τι, τι σημαίνει αυτό. Δεν προκύπτει νομίζω από το κείμενο και τέλος οι τυποποιημένες διαδικασίες ακούγεται καλό αλλά δεν είναι καλύτερο να έχουμε καλά δίκτυα για να μην προσαρμόζονται διάφορες διαδικασίες και πρωτόκολλα. Νομίζω πως αυτό λειτουργεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ιδανικά εγώ θα ήθελα να σταματήσει να εφαρμόζεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να είμαι ρεαλιστής και να μιλήσω καλύτερα για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές πρώτα απ' όλα τα ε, δικαστήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να πισθούν πέραν αμφιβολίας ότι υφίσταται η βάση, νομική βάση για την ποινική δίωξη τώρα θα δοθεί η δυνατότητα απόρριψης του εντάλματος με βάση ανησυχίες ανθρωπινών δικαιωμάτων. Εμείς θα επιθυμούσαμε να υπάρχει η υποχρέωση από το ε, κράτος μέλος που εκδίδει το ένταλμα σύλληψης να ε, υποβάλει και να υποδεικνύει και τεκμήρια. Η κυρία Λάτφορτ, αν κατάλαβα καλά, αναφέρθηκε στην χρήση του εντάλματος αυτού για την προσαγωγή μαρτύρων και όχι υπόπτων. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια κατάχρηση του εντάλματος και κατά πάσα πιθανότητα τα κράτη που το έκαναν αυτό το έκαναν εν γνώση τους και αναρωτιέμαι ποιες θα είναι οι συνέπειες που θα υποστούν. Επίσης αναφέρατε, κυρία Συγήτρια, ότι πολλές φορές το ένταλμα χρησιμοποιείται ω η πρώτη επιλογή αντί για την τελευταία επιλογή. Θα πρέπει να απορρίπτεται σε εκείνε τις περιπτώσει. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ε, διαφορετικό όταν κάποιος ε, εκδίδεται από τη χώρα του προς άλλη χώρα και διαφορετικό όταν από τρίτη χώρα επιστρέφει στη χώρα του για να δικαστεί. Ακούσαμε τον κύριο Μέλο ότι υπήρξε συμφωνία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα έρευνα. Κανονικά ούτε υπέρ αυτού του εργαλείου θα ήμουν, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης θα προτιμούσα πριν τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ένταλματος Σύλληψης να χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα έρευνα τουλάχιστον. Γιατί διαφορετικά ε, δεν γίνεται σωστή ε, δίωξη ε, υποθέσεων. Επίση διάβασα ότι μόνο 11.500 1.500 εντάλματα σύλληψη τελικά εκτελέστηκαν, ενώ ήταν πολύ περισσότερα εκείνα τα οποία αιτήθηκαν. Και αναρωτιέμαι γιατί συνέβη αυτό. Ναι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την γνωμοδότηση. Μια και πρόκειται να ε, ενημερωθούμε και μια σειρά νέο μέτρο που προετοιμάζει η Επιτροπή στον τομέα αυτό. στον τομέα της ποινικής συνεργασίας χρειάζεται μια ε, συνεργασία σε, σε, σε, μεταξύ κρατών μελών γιατί η κλιματικότητα είναι διασυνοριακή και ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα το θεωρώ επιτυχημένο προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνώ επίσης με τον συνάδελφο που είπε ότι τα προβλήματα έγκυται στην εφαρμογή. Πριν εκλεγώ μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπούσα την κυβέρνηση της Μάλτας το Συμβούλιο Δικαιοσύνης ε, και Ιστορικών Υποθέσεων και θα ήθελα να σας πω ότι η συζήτησή μας στην ομάδα ΔΕΗ κατά κύριο λόγο αναφερόταν στον αναλογικότητα και στον τρόπο εφαρμογής αυτών των εργαλείων. Και επίσης τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των ορισμών των αξιόπινων πράξεων από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόβλεψη για έλεγχο αναλογικότητας, καθώς επίσης και το ζήτημα των ενδικών μέσων, στα οποία αναφέρθηκε και ο κ. Κέρκορπ. Πολύ συχνά συναντούμε ε, θύματα στις χώρες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την απονομή δικαιοσύνης που θα άξιζαν τελευταίο σημείο και ερώτημα προς την εισηγήτρια, ενώ μιας πιο αναλυτικής ε, συζήτησης στο μέλλον. Νομίζω ότι δεν είναι ο στόχος μας εδώ να ζητήσουμε πλήρη αναθεώρηση της απόφασης πλαίσιο. Ιδίως όσον μιας και τώρα ε, ετέθησε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνα. θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στο μέλλον. Και τώρα η Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την γραμμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση αξιολόγηση του 2011, τα ευρήματα της οποίας συνεχίζουν να, ε, είναι, ισχύουν, το ζήτημα της αναλογικότητας είναι το πιο σημαντικό, καθώς επίσης και το θέμα των στατιστικών στοιχείων της εκπαίδευσης και η βελτίωση του σεβασμού των δικονομικών ε, δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Θεωρούμε ότι, υπάρχει καλή, ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης λειτουργεί ε, καλά και έχει βοηθήσει την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και προτείνει ε, βελτιώσεις στον τομέα των δικονομικών δικαιωμάτων οι οποίες βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πρόσφατα εγκρίθηκε η οδηγία ε, για την πρόσβαση σε δικηγόρο, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον κατηγορούμενο να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο και στις δύο χώρες. Σήμερα η Επιτροπή θα εγκρίνει μια νέα σειρά ε, ε, πρωτοβουλειών για τα δικονομικά δικαιώματα, ανάμεσα σε αυτές μια πρωτοβουλία για την δωρεάν νομική συνδρομή, το Legal Aid, υπάρχουν και άλλα εργαλεία ποινικής συνεργασίας, όπως για παράδειγμα η απόφαση πλαίσιο για την επιτήρηση. Αυτά θα μπορούσαν, όπως είπε και η συγγήτρια, να συνεισφέρουν και να ε, μειωθεί η ε, προφυλάκηση στα κράτη-μέλη. Τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε η κατάσταση, κυρίως σε σχέση με το ζήτημα της αναλογικότητας. Εδώ έχουμε σαφή βελτίωση όλο και λιγότερες είναι, τα αιτήματα ε, χωρίς βάση. Από το 2014 και μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει αρμοδιότητα ελέγχου αυτών των ε, ενταλμάτων και αυτό θα αλλάξει τα πράγματα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί βέβαια τις εξελίξεις και μετά την υιοθέτηση της ε, γνωμοδότησης από την Επιτροπή ε, του Κοινοβουλίου, τη ΛΥΜΠΕ, θα την εξετάσουμε η Πρόεδρος αναρωτιέται. Μάλλον δεν θέλει να επανέλθει η Προεδρία, επομένως κύριε Λάτφορντ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη στήριξη των ασκείωδων εισηγητών. Είμαστε, θα έλεγα, μια ομάδα που εργάζεται σε όλα τα ζητήματα ποινικού δικαίου και υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία συναδέλφους. Η κυρία Σίπελ ήταν η συγγήτρια της οδηγίας για το δικαίωμα σε δικηγόρο που αναφέρθηκε και νομίζω πως το Κοινοβούλιο έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων π.χ. το να υπάρχει παρουσία δικηγόρου και στο κράτος που εκδίδει το ένταλμα. Εμείς πιέσαμε γι' αυτό όπως ε, και στο Ευρωπαϊκό Εντάλμα Έρευνας. εμείς ζητήσαμε να υπάρχει απόρριψη λόγω θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και θα έλεγα μάλιστα πως ε, εάν είχαμε συναπόφαση το 2002 θα είχαμε καλύτερο ένταλμα και γρηγορότερες διαδικασίες όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα γιατί το κενό των 9 ετών μεταξύ του εντάλματος και των πρώτων μέτρων ε, δικονομικού χαρακτήρα ήταν ε, ακριβώ πάρα πολύ μεγάλο. Πράγματι, έχετε δίκιο λοιπόν, ασχολούμαστε με προβλήματα που υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία και θα τα είχαμε λύσει, δεν θα ήμασταν τώρα σε αυτή τη θέση. Καλοδεχόμενη λοιπόν η στήριξη ε, όλων όσων μίλησαν. Δεν ζητάμε να καταργήσουμε το ένταλμα απλά να το βελτιώσουμε. Να πω κάτι στον κύριο Ντε Στην παράγραφο 1 λέμε, λέμε πως δεν θα πρέπει να ασχοληθεί η έκθεση με προβλήματα που προκύπτουν αμέσως, άμεσα από την ε, μη τήρηση των κανόνων. Δηλαδή εδώ πρέπει να μιλάω για τις προθεσμίες. Όταν ε, πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα τα κράτη-μέλη όπως αναγράφονται στο ένταλμα και δεν ε, τα κάνουν. Ε, αυτό δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία. Για τέτοια ζητήματα λοιπόν μιλάω. Γεγονός είναι πως το σχέδιο αυτό έκθεσης δεν ορίζει το εάν οι νομοθετικές λύσεις ε, που ζητάμε θα πρέπει να είναι να ξαναγραφτεί η σχετική απόφαση ή άλλα μέτρα πιο οριζόντια που θα αφορούν όλα τα μέσα αμοιβιάς αναγνώρισης. Αυτό λόγω και έλλειψης ε, βεβαίως χώρου αλλά και γιατί ε, μερικοί συνάδελφοι το ανέφεραν, υπάρχει και το ζήτημα του κουτιού της Πανδώρας. Δηλαδή, εάν το ανοίξουμε το ζήτημα θα έχουμε καλύτερη λύση ή θα έχουμε ε, οπισθοδρόμηση και θα πάμε στο παλαιό σύστημα έκδοσης. Και βεβαίως θα επιτρέψει σε κάποια μέλη που δεν θα κατανομάσω πάρουν απόφαση για το εάν ε, θα επανενταχθούν σε ένα νέο ένταλμα. Εγώ δεν θέλω να ξαναπεράσουμε αυτή τη διαδικασία. Και το κομμάτι ακριβώς ε, της ε, νοοθικής μεταρρύθμισης το έχω αφήσει αμφίσιμο Μπορεί οι συνάδελφοι να θέλουν να το αλλάξουν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να τονίσουμε τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα θέματα και όχι τον τρόπο. Κατόπιν, κύριε Τάου, η πρόταση νομικής ε, αρρωγής αφορά την παροχή αυτή στην αρχή της ποινική διαδικασίας. Δεν ξέρω τι λέει αυτό. Ε, γιατί νομίζω υπάρχει μια σύσταση για τις υπόλοιπες περιπτώσεις και οπωσδήποτε θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και σχόλια. προσωπική μου άποψη βεβαίω είναι πως θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται με τις ε, συνθήκες ε, κράτησης που είναι σοβαρό ζήτημα στην ε, εφαρμογή του εντάλματος αυτού γιατί βεβαίως δεν θα πρέπει να προφυλακίζονται οι άνθρωποι για χρόνια και σε κακές συνθήκες. Τέλος. Οι δύο πανεπιστημιακοί, οι δύο ειδικοί κάνουν κάποιες εκθέσεις ε, στην μονάδα ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας προετοιμάζουν τις εκθέσεις τους. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τους συναντήσουμε. Να τους συναντήσουν οι σκιοδεσηγητές, δηλαδή την κυρία Ντιουμπέ και τον κύριο Βέρνερ. Αναμένουμε το σχέδιο των εκθέσεών τους σε προσεχές μέλλον. Αλλά ήδη έχουμε κερδίσει από τις ε, πρώτες ε, σκέψεις τους ε, που ενσωματώθηκαν στην έκθεση. Ο κύριος Κέκχοπ είπε πως θέλουμε να γίνουν αυτά τα οποία ζητάμε. Πράγματι, οι συγητές και οι έχουν αυτή την άποψη. Θέλουμε να γίνουν αυτές οι αλλαγές και αν επανεκλεγούμε θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία και βεβαίως πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να κάνει κάτι αλλά υπάρχει Βεβαίω η δυνατότητα να κάνει κάτι μια ομάδα κρατών Αν δεν μπορεί ή δεν θέλει η Κομισιόν θα πρέπει να το συζητήσουμε ίσως με κάποια κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν πως υπάρχει διάθεση να λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης με τρόπο αποτελεσματικό και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλιώς βλάπτεται η φήμη του και θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε απολογία. Πρέπει να γίνουν λοιπόν αυτές οι αλλαγές και η Κομισιόν πρέπει να ακούσει το Κοινοβούλιο εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Βαρόνι Λάτφορτ όπως είπατε οι προθεσμοί για τροπολογίες ε, είναι μόλις στις 6 Δεκεμβρίου. Τελειώνουμε με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και περνάμε στις ψηφοφορίες σε δύο λεπτά. Οπότε, όποιος θέλει να φύγει από την αίθουσα παρακαλώ τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όποιος δεν επιθυμεί να ψηφίσει, ας ε, βγει από την αίθουσα. Και να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Δύο θέματα έχουμε. Σφυράκι. Χρησιμεύει καλύτερα το σφυράκι εδώ. Δύο ψηφοφορίες στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα το, θέμα, το πρόγραμμα Περικλής 2020 για την ανταλλαγή, συνδρομή και κατάρτιση για την προστασία του ευρώ από την παραχάρεξη και την κινδυλία. Υπάρχει συμφωνία με το Συμβούλιο και ο εισηγητής προτείνει να υπερψηφίσουμε ομού το συμβαστικό κείμενο. Κύριε Μάκιντάρ, θέλετε το λόγο μήπω. Κύριε Μάκιντάρ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω και πολλά. Θέλω απλώ να ευχαριστήσω όλου του χειώτε συζητητέ σε αυτό το φάκελο και αυτό το φάκελο. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε, γιατί ε, προβλεπόταν ότι το πρόγραμμα Περικλή 2020 θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Ε, Επομένω, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει συμφωνία. Όλοι, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, οι σκιώδει το υποστηρίζουν. Ευελπιστώ λοιπόν ότι θα το υπερψηφίσουμε και θα προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε. Προτείνω λοιπόν να τεθεί στη ψηφοφορία το σύνολο του ε, συμβιβαστικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι σαφές λοιπόν ότι εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά όμως αυτή τη φορά. Έναρξη ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορία. Ομόφωνα υπέρ. Συγχαρητήρια κύριε Μάκιντρα. Εγκρίνεται. Κύριε Μακίντερ, να προσθέσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων προς όλους τους συναδέλφους. Μήπως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας το Δεκέμβριο. Θα ήταν σκόπιμο να μην καθυστερήσει το πρόγραμμα. Οι πρόεδρος μου είπαν ότι υπάρχει το ζήτημα με τους γλωσσομαθείς νομικούς που θα πρέπει να εξετάσουν το κείμενο. Θα το προσπαθήσουμε πάντως. Ευχαριστούμε κυρία Μάκιντάι. Όπως είπα το πρωί, τα σημεία 8 και 9 ε, τους διάταξης έχουν αναβληθεί. Επομένως απομένει το σημείο 10. Κατάγερση της απόφασης 2007-124 ε, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Βρατών. Οι συντονιστές στις 17 ε, Σεπτεμβρίου αποφάσισε να ακολουθηθεί η απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 46. Επομένω, προχωράμε αμέσω στην ψηφοφορία. Ε, μία και μοναδική ψηφοφορία επί τη ε, προσχεδίου γνωμοδότηση. Δεν υπάρχουν τροπολογίε υπέρ. Όχι, με ενημερώνει η γραμματεία ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικά αυτή την ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία ηλεκτρονική, παρακαλώ. Κλήξη. 37 υπέρ, Δύο κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο ως τροποποιήθηκε. Όχι, δεν χρειάζεται. Το κάναμε ήδη. Ωραία, άρα ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες για σήμερα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Και προχωράμε στο σημείο 11 της μερικής διάταξης. Παρακαλώ συνάδελφοι, όσοι φεύγουν από την αίθουσα, ας το πράξουν για να συνεχίσουμε. We're going to ask the speaker, which is the, the, the, the Uh, Συναδελφοί, το ζήτημα των αγνοωμένων στην Κύπρο έχει αποτελέσει διαχρονικά ζήτημα ανησυχίας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Έχουμε εγκρίνει ε, ψηφίσματα το 2007 και το 2008, καθώς επίσης και μια δήλωση του Κοινοβουλίου του 2011. Πέρυσι το Δεκέμβριο μια αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών με πρόεδρο, ε, τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ, επισκέφθηκε την Κύπρο και είχε τη δυνατότητα να ε, έχει ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Προσφύγων Εγκλωβισμένων και Αγνοημένων και παθόντων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας της ε, Κύπρου. Η πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, η κυρία Σκέβη Κουκουμακούτρα, βρίσκεται εδώ σήμερα. Οι συντονιστές της Επιτροπής Λίβε ε, αποφάσισαν να την προσκαλέσουν, την κυρία Κουκουμακούτρα, να, για να μας ενημερώσει ε, για το, την κατάσταση όσον αφορά αυτό το σημαντικό ανθρωπιστικό ζήτημα. Κυρία Κούτρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή στο σύνολό τη για τη δυνατότητα να ενημερώσουμε για το θέμα των αγνωμένων και των τελευταίων εξελιξιών. Όπως ξέρετε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 άφησε πίσω πρόσφυγες, νεκρούς, τραυματίες αλλά και εκατοντάδες αγνοούμενους. Νεκρούς και αγνοούμενους άφησαν πίσω τους και οι συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που διαπράχθησαν από το εθνικιστικό μίσος κυρίως κατά τη δεκαετία του 60. Ο αριθμός των αγνοωμένων της Κύπρου είναι 1508 Ελληνοκύπριοι και 493 Τουρκοκύπριοι. Τον Απρίλιο του 1981 συστάθηκε η διαρευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αποστολή της είναι η διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων της Κύπρου. Η διαρευνητικη Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη. Έναν εκπρόσωπο της ελληνοκυπριακής πλευράς, έναν εκπρόσωπο της τουρκοκυπριακής πλευράς οι οποίοι επιλέγονται από τις δύο κοινότητες αντίστοιχα και το τρίτο μέλος το οποίο επιλέγεται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα τα τρία μέλη της ΔΕΑ είναι ο κύριος Θεοφίλου, εκ μέρου της ελληνοκυπριακής κοινότητας, η κυρία Κουτσούκ, εκ μέρου της τουρκοκυπριακής κοινότητας και ο κύριος Πολ Χένρι Αρνή, το τρίτο μέλος διορισμένος από τα Ηνωμένα Έθνη. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί με τη μέθοδο του DNA τα οστά 456 αγνοωμένων. Οι 358 από αυτούς είναι Ελληνοκύπριοι και οι 101 Τουρκοκύπριοι. Σήμερα εργάζονται 9 συνεργεία εκταφών στις κατεχόμενες περιοχές και 3 συνεργεία στις ελεύθερες περιοχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανθρωπολογικό εργαστήριο έχει στελεχωθεί με επιπλέον επιστήμονες όπως γενετιστές, ανθρωπολόγους και τη συντονίστρια ταυτοποιήσεων. Είναι γεγονός ότι ο χρόνος λειτουργεί αρνητικά για το ζήτημα των αγνοωμένων. Για τον λόγο αυτόν η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε δημόσια ανέκκληση πρόσφατα σε όσους έχουν πληροφορίες αναφορικά με αγνοούμενους και σημεία ταφής αγνοωμένων να τις δώσουν το συντομότερο. Μέσα από τα αναλυτικά στοιχεία που δίνει η Διαρευνητική Επιτροπή διαφαίνεται η ανάγκη για εντατικοποίηση της προσπάθειας για συλλογή πληροφοριών γιατί ο χρόνος είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας των τομέων αυτών. Σαράντα χρόνια μετά σημαντικοί μάρτυρες έχουν αποβιώσει ή ακόμα και τα σημεία ταφής αγνωμένων που θυμούνται αυτόπτες μάρτυρες να έχουν αλλοιωθεί από το χρόνο. Αυτό δυσκολεύει τις εργασίες εκταφής διότι συχνά των τελευταίων καιρών οι εργασίες αυτές δεν οδηγούν στον εντοπισμό λιψάνων. Σύμφωνα με τη Διερευνητική Επιτροπή, από τα 797 σημεία εκταφών που πραγματοποιήθηκαν από το 2006 μέχρι σήμερα, μόνο στα 271 σημεία εντοπίστηκαν λείψανα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπολογίζεται ότι υπάρχουν ακόμα περίπου 300 σημεία που πιθανότατα υπάρχουν θαμμένοι αγνοούμενοι και από αυτά τα 30 σημεία είναι σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από τον τουρκικό στρατό ως στρατιωτικές περιοχές. Είναι γνωστό βέβαια ότι οι τοποθεσίες όπου υπάρχουν ομαδικοί τάφοι έχουν κηρυχθεί από τον τουρκικό στρατό ως στρατιωτικές ζώνες για να μην είναι προσπελάσιμοι στο κοινό. Γι' αυτό ζητούμε όπως ασκηθεί περαιτέρω πίεση στην Τουρκία για να επιτρέψει την πρόσβαση σε στρατιωτικές περιοχές για να γίνουν εκταφές. Επιπλέον ζητούμε όπως δοθούν στοιχεία μέσα από τα αρχεία του στρατού της Τουρκίας. Υπάρχουν πληροφορίες τις οποίες κατέχει η Τουρκία και ο κατοχικός στρατός, οι οποίες δεν έχουν δοθεί, πράγμα που αποδεικνύεται και με την πρόσφατη δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως και περιέχει σκηνές από μεταφορά εχμαλώτων του 1974. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιστήμονες της Διερευνητικής Επιτροπής διαπιστώνουν ότι υπήρξε μετακίνηση οστών, έργων που σίγουρα έχει εκτελέσει ο κατοχικός στρατός. Και να πω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν δημοσιευθεί σε εφημερίδες πληροφορίες ότι το 1996 με μια εκστρατεία από την Τουρκία είχα γίνει εκταφές οστών και είχαν, λένε οι πληροφορίες, πεταχτεί στη θάλασσα. Αν η Τουρκία δώσει πληροφορίες, τότε το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Το άρθρο 11 των όρων εντολής της Διερευνητικής Επιτροπής, όπου αναφέρεται ότι η διερευνητική δεν θα επιχειρήσει να αποδώσει ευθύνη για το θάνατο οποιοδήποτε αγνοούμενου ή να ερευνήσει την αιτία τέτοιων θανάτων. Θα έπρεπε να ρυθμιστεί και διασυνδεθεί με την ετοιμότητα να δοθούν πληροφορίες για τη διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων και όχι μεγάλο μέρος των εργασιών, όπως είπα πιο πάνω, να είναι, αναπο... αναποτελεσματικών και να μην οδηγεί στον εντοπισμό λιψάνων. Πάγιον αίτημα προς, αυτήν την κατεύθυνση των συγγενών των αγνοωμένων είναι και η εξυχνίαση των συνθηκών που χάθηκαν οι δικοί τους και η απόδοση ευθυνών, θέμα για το οποίο διεθνείς θεσμοί προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να σταθούν στο πλάι τους. Με την αύξηση του αριθμού των ταυτοποιήσεων έχει διαφανεί επίση η αναγκαιότητα ρύθμιση τη έκδοση των πιστοποιητικών θανάτου που δίνονται στου συγγενείς των αγνωμένων που έχουν ταυτοποιηθεί τα οστά και έχουν κυδευθεί. Όπω φαίνεται στα πιστοποιητικά θανάτου, αναγράφεται ω άγνωστη η αιτία θανάτου. Και έχω μαζί μου μερικά τέτοια πιστοποιητικά θανάτου που πραγματικά προκαλούν συγκλονισμό. Ο Νίκος Εγκλέζος, που έχουν ταυτοποιηθεί τα οστά του, στο πιστοποιητικό θανάτου αναφέρει άγνωστη αιτία και πιο κάτω περιγράφει ότι ε, είχαν εντοπιστεί στον Νίκο τρία τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, τραύμα από σφαίρα στον αριστερό μυρό, στον αδελφό του τραύματα από σφαίρα στο κρανίο, στα πόδια, στο θώρακα, το ίδιο στον πατέρα τραύμα σφαίρα στο δεξιό μυρών στις πλευρές. Τέτοια πιστοποιητικά, τέτοιες περιγραφές νομίζω ότι αδικούν την έκδοση πιστοποιητικών θανάτων που να παραπέμπουν σε άγνωστη αιτία θανάτου. Αν λοιπόν θεωρώ ότι είναι θέμα ηθικής υποχρέωσης προς τους συγγενείς των ελλονοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αγνοωμένων, αλλά και ιστορικής μνήμης να αναφέρεται στα πιστοποιητικά θανάτου των αγνοωμένων, των ότι η ταυτότητα τους διαπιστώθηκε με αναλύσεις με τη μέθοδο DNA, παραδείγματο χάρη, ότι ο ταυτοποιητής ήταν αγνοούμενος από τον πόλεμο του 1974 ή των διακοινωτικών του 1963-1964 και ότι τα οστά του εντοπίστηκαν σε τάφον σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Θεωρώ επίση ότι τα πιστοποιητικά θανάτου θα πρέπει να εκδίδονται από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνωμένων, αφού είναι στα πλαίσια του δικού τη προγράμματο που έγινε ο εντοπισμό και η ταυτοποίηση των οστών. Όσον αφορά τον προπολογισμό τη Διερευνητική Επιτροπή, πέραν από το κονδύλι 2,6 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εργασίε που επιτελεί η ε, διαρευνητική Επιτροπή και αφορούν τον προπολογισμό του 2014, η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλει προσπάθειες για να εξεύρει και άλλους δωρητές, αφού υπάρχει ήδη έλλειμμα 500.000. Από τον Ιούνιο του 2012 έχουν ξεπεραστεί κάποια προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια και η αγαστή συνεργασία της ΔΕΑ με, το διεθνές, με τη Διεθνή Επιτροπή Αγνοουμένων δίνει τη δυνατότητα εντατικοποίηση των εργασιών του προγράμματο ταυτοποίησεων. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι από το 2006 μέχρι το 2013 έχει εισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ταμείο αυτών 12.718.000 η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εισφέρει 3.183.000 η Τουρκία 637.000 και κάποιες άλλες χώρες όπως παραδείγματος χάρη η Αγγλία 220.000, η Γερμανία 263 και άλλες με μικρότερα ποσά τις, τις οποίες θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συμβολή αυτή. Θεωρούμε όμως σημαντικό αυτή τη στιγμή να στηριχθεί ακόμα περισσότερο οικονομικά το πρόγραμμα ταυτοποίησης αφού μπορούν να εντατικοποιηθούν περισσότερο οι εργασίε του. Ζητούμε τη δραστική επίση παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να στηριχθεί το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής. Ζητούμε τη συμβολή σας ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και να συμβάλλει στην εξακρίβωση της τύχης των αγνωμένων. Οι οικογένειες των αγνωμένων έχουν κάθε δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια για τις συνθήκε υπό, υπό τις έχασαν τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια τους. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι σε έναν πολύ μικρό νησί όπως η Κύπρος με πληθυσμό κάπου στο έναν εκατομμύριο, ο χρόνος δεν επουλώνει τις πληγές. Μόνον η αλήθεια επουλώνει τις πληγές. Και η επίλυση του ζητήματος των αγνοωμένων είναι πρώτη στα έναν ανθρωπιστικό ζήτημα. Είναι όμως και μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η Κύπρος να ξεκολλήσει από το παρελθόν και να γυρίσει τη σελίδα του μέλλοντος. Με τον λαό της ενωμένο, με τη γη μας ελεύθερη και απαλλαγμένη από στρατούς και σειρματοπλέγματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και τη δυνατότητα να κάνω αυτή την παρουσίαση. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις αν υπάρχουν. Thank Σας ευχαριστούμε. Πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ε, καλά κάνατε και ήρθατε και μας ε, ενημερώσατε. Ε, υπάρχει κάποιο που θα ήθελε να παρέμβει. Ναι, ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο Πρόεδρο της Αρμόδιας Επιτροπής από το Κυπριακό Κοινοβούλιο για την παρουσίαση της. Έχω εντοπίσει τρία-τέσσερα σημεία που θα ήθελα να θίξω και είναι σημεία τα οποία ως αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που επισκεφθήκαμε τον περασμένο Δεκέμβριο την ε, Κύπρο τα είχαμε εντοπίσει και τότε και το πρώτο είναι η απέτηση για πρόσβαση στις ε, στρατιωτικές περιοχές. Ε, νομίζω ότι είναι χρόνος πλέον να απαιτήσουμε ως Κοινοβούλιο από τις ε, τουρκικές αρχές, ιδιαίτερα τις στρατιωτικές, να βοηθήσουν έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επισκεφθεί, η Επιτροπή Αγνωμένων εννοώ, ε, αυτές τις περιοχές και να κάνει τις έρευνες οι οποίες χρειάζονται διότι εκεί είναι που υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν λήψη αναγνωμένων. Το άνοιγμα των αρχείων των στρατιωτικών αρχών είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό διότι εκεί υπάρχουν οι πληροφορίες Τώρα έχουν περάσει 40 χρόνια από την εισβολή και οι δικαιολογίες που εδίδονται στο παρελθόν νομίζω ότι τώρα έχουν εκλείψει ε, και θα μπορούσε το Κοινοβούλιο μας να βάλει ε, πίεση πάνω στις ε, αρχές της Τουρκίας για να ανοίξει αυτά τα αρχεία. Το τρίτο σημείο που έχει λεχθεί και νομίζω είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα των πιστοποιητικών θανάτου είναι λίγο παράδοξο να βλέπει ένας ένα κρανίο με μία τρύπα στο μέτωπο και να λέει άγνωστη αιτία θανάτου. Τουλάχιστον θα έπρεπε ένα πιστοποιητικό να συνάδει με τα πραγματικά ευρήματα σε ό,τι αφορά τα λείψανα που εντοπίζονται. Τέταρτο σημείο είναι αυτό του προϋπολογισμού Έχουμε κάνει κάποιες τροπολογίες στον περασμένο προϋπολογισμό για να βοηθήσουμε, αλλά αυτό το έλλειμμα των 500.000 νομίζω ότι ε, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να προσπαθήσουμε και με ε, donations από τα κράτη-μέλη, αλλά επίσης από τον προϋπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλυφθεί. Και τέλος θέλω να πω κάτι το οποίο είχα πει και σε προηγούμενες ε, συνεδρίες της Επιτροπής μας, χωρίς όμως ε, να το έχουμε παρακολουθήσει. Το 2008 ε, στην έκθεση της Επιτροπής μας με εισηγήτρια την κυρία Κλάμπτ τότε, στο σημείο 6 είχαμε πει ότι η Request the Committee on Civil Liberties έλεγε αυτή η έκθεση to follow up the issue of missing persons in Cyprus and to submit annual reports. We haven't, Madam Chair, done this. We have not, as a Civil Liberties Committee, η Επιτροπή Θελειοδών Ελευθεριών δεν το έκανε αυτό. Το, την, ε, θυμάμαι τη συνάδελφα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά έφυγε νομίζω το 2009 και μετά αποφασίσαμε ο κύριος ε, Μπουσουτήλ να είναι ο εισηγητής που θα την διαδεχόταν όπως και έγινε αλλά και αυτός έφυγε χωρίς να υποβάλει ετήσια έκθεση και τώρα έχουμε μείνει χωρίς εισηγητή. Προτείνω λοιπόν να θέσουμε αυτό το ζήτημα στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών για να αποφασίσουμε το εάν θα πρέπει και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εισηγητή για το ζήτημα των αγνοωμένων. Σας ευχαριστώ. Thank you. I do agree with you and σας ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη πως η επόμενη συνεδρία των συντονιστών θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Σίγουρη. Θα δούμε λοιπόν τι θα πούν οι συντονιστές. Η κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι οι κυβερνήσει στην Κύπρο βλέπουν το θέμα των αγνωμένων ως καθαρά ανθρωπιστικό θέμα και για πολλά χρόνια τώρα το συζητούν σε διεθνή βήματα και είναι γεγονός ότι υπάρχουν σχετικά ψηφίσματα και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κρίμα γιατί αναγκαζόμαστε μετά από 39 χρόνια να συζητούμε ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα όλα αυτά τα χρόνια γιατί είναι αναφέρει το δικαίωμα των συγγενών να γνωρίζουν τι απέγιναν οι δικοί τους, τα δικά τους άτομα. Ε, θα πω ότι σε επισκέψεις που έχουμε πραγματοποιήσει και ως Ευρωβουλευτές και με την παρουσία άλλων συναδέλφων στο εργαστήριο διακρύβωσης της τύχης των αγρομένων στη Λευκοσία ήταν πάντα εφανές ότι αρκετά από τα κρανία που εκείτοντας τα τραπέζια εκεί μας τα είχαν δείξει οι εμπειρογνώμονες που ήταν και ελληνο και Τουρκοκύπροι είχαν στο σημείο του μετόπου μία τρύπα και δυστυχώς οι όροι εντολής της Δερευνητική Επιτροπής δεν επιτρέπουν να γίνει και ξυχνίαση των αιτίων του θανάτου. Και αυτό είναι τραγικό, γιατί όταν δίνεις τη σωρό μετά τη διακρύβωση με τον DNA στους συγγενείς και το, πιστικό, το πιστοποιητικό γράφει αιτία θανάτου άγνωστη, Δικαιολογημένα οι συγγενείς διερωτούνται «Καλά, αυτή η τρύπα στο κρανίο τι ήταν» και όταν υπάρχουν ευφανείς σημάδια για πυροβολισμούς σε διάφορα σημεία του κορμιού, αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται και είναι πολύ εύλογη ανησυχία γιατί γράφεται αιτία θανάτου άγνωστη όταν γνωρίζουμε ότι αυτά τα παιδιά, κυρίως 18-19 χρονών, οι πλήστοι από αυτούς ήταν στρατιώτες που αντιμετώπισαν την τουρκική εισβολή. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να δούμε αν στο μέλλον επιβάλλεται ο όρος εντολής της δερευνητικής να αυξηθεί για να μπορεί πραγματικά να μην γράφει αυτόν τον τραγελαφικό αιτία θανάτου άγνωστη. Όμως για να είμαστε πρακτικοί, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ανησύγηση στη δική μας Επιτροπή, γιατί γνωρίζετε κάθε χρόνο εδώ εξετάζεται η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Και η έκκληση μου είναι αυτή η Επιτροπή που ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα, πραγματικά στην έκθεση πρόοδου της Τουρκίας να ασκηθεί πίεση και να γραφτεί κάτω υπό μορφή τροπολογιών. Ίσως η Επιτροπή θα μπορούσε να το προωθήσει ότι η νέη Τουρκία πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε στρατιωτικές περιοχές γιατί υπάρχουν στην Κύπρο και υπάρχουν και σε άλλες περιοχές εκτός Κύπρου όπου υπάρχουν ε, στοιχεία ότι πιθανόν να βρίσκονται Κύπροι αγνώμενοι και δυστυχώς κάθε φορά που εντοπίζεται μια στρατιωτική περιοχή η, το ψευδοκράτος απαγορεύει την πρόσβαση και κηρύσσει νέες στρατιωτικές περιοχές που είναι λάθος. Αυτό παρακολεί το έργο της Διευνητικής Επιτροπής. Και επίση η πρόσβαση στα στρατιωτικά αρχεία. Θυμούμαι όταν ήμουν μέλο του Συμβουλίου τη Ευρώπη, περάσαμε motions, resolutions και εζητήτων από την Τουρκία να ανοίξει τα στρατιωτικά αρχεία στη Δερευνητική Επιτροπή. Δεν το έχει πράξει. Αν δεν ασκηθούν πιέσει στην κατοχική πλευρά που είναι η Τουρκία, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε για αυτό το θέμα, το συζητούμε ακόμα 50 χρόνια. Θα πεθάνουν οι συγγενείς και δεν θα μάθουν τι απέγιναν οι δικοί τους. Και το τελευταίο, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Για μένα είναι αδιανόητο η Τουρκία ως υποψήφια για ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει κάθε χρόνο εκατομμύρια ε, χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια στα οποία η χώρα μου η Κύπρος συμμετέχει ως ε, χώρα donor country. Είναι αδιανόητο η Τουρκία να παρέχει μόνο 630.000 ευρώ όταν παίρνει πέραν των 900 εκατομμυρίων ετήσια. Και διερωτούμε, δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφαιρεί έναν ποσό για να χρηματοδοτείται η προσπάθεια διακρύβωσης αυτών ακριβώς των ατόμων που δυστυχώς εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι λόγω της υπετιότητας της Τουρκίας και τη τουρκικής εισβολής του 1974. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Κύριος Κλέης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω 100% με τους δύο Κύπριους συναδέλφους. Επιτέλους, δεν είναι δυνατόν το 2013 να συζητάμε στην Επιτροπή μας για το πρόβλημα των αγνοωμένων όταν έχουμε την ε, κολυσιεργία της ε, Τουρκίας ε, για να μην διαπιστώσουμε πού βρίσκονται οι άνθρωποι και υπό ποιες συνθήκες πέθαναν. Να σκεφτούμε πως ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2005 και όλον αυτό τον καιρό ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος σε αυτό το ζήτημα και σε πολλά άλλα. Βεβαίως που είναι εξίσου σημαντικά, σκεφτούμε την άρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει σε πλοία και αεροπλάνα ε, κυπριακά να πάνε σε τουρκικούς λιμένες και αερολιμένες με όλα αυτά πραγματικά δείχνουν και την ασθενή διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ασκεί καμία πίεση για αρνείται να ασκήσει και δεν πρέπει να μας προξενεί έκπληξη το ότι δεν έχει σημειωθεί άρα καμία πρόοδος. Είναι πραγματικά έσχος το ότι πρέπει σήμερα να ζητάμε, ε, να παρακαλάμε τις ε, τουρκικές αρχές για συνεργασία. Αυτό από μόνο του θεωρώ πως είναι αιτία να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε ξανά στην ε, κυρία Κουκουμά Κούτρα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να ευχαριστήσω όσους πήραν τον λόγο. Σίγουρα τους δύο Κύπριους Ευρωβουλευτές για τις παρατηρήσεις ε, που με, την, ε, με τις διευκρινήσεις που έχουν κάνει νομίζω έχουν κάνει πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πώς η αδικία γίνεται σε αυτή την περίπτωση αλλά σίγουρα να συμφωνήσω και με τον κύριο Κλέη για το πώς στεκόμαστε απέναντι στην Τουρκία το πώς ανεχόμαστε τη δική της στάση και συμπεριφορά ακόμα και εκεί που έχει ευθύνες τις οποίες έχουν όλοι ε, παραδεχτεί και τις υποδεικνύουν με πάρα πολλά ψηφίσματα σε διάφορα επίπεδα από τα Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και να έρθουμε σε περιφερειακούς θεσμούς και οργανισμούς, τα οποία στην Κυπριακή λέμε ότι γράφει στα παλιά τη τα παπούτσα και δεν σέβεται με κανέναν τρόπο. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και οι άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν διαφορετικό ρόλο, να ασκήσουν τις πιέσεις ε, ακόμα πιο έντονα και σε σχέση με την ένταξη της Τουρκίας ε, και τις διαδικασίες και δεν μπορεί να ανεχόμαστε ε, αυτή τη συμπεριφορά. Το πώς είχε συμπεριφερθεί, παραδείγματο χάρη, στα, όταν, η Κυπριακή, όταν Κύπρος ασκούσε την ε, Προεδρία του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω καταδεικνύει με ποιον τρόπο να αντιμετωπίζει ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους θεσμούς. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε όχι μόνο δεν σεβάστηκε την Κύπρο που ασκούσε την Κυπριακή Προεδρία, αλλά είχε καλέσει και άλλες χώρες να μην συνεργαστούν ακριβώς στα πλαίσια εκείνα. Ε, νομίζω σύστατη προσπάθεια και τελευταίο μου σχόλιο είναι τη δική σας συμβολή, τη δική σας συμπαράσταση στους συγγενείς των αγνοωμένων που για 40 χρόνια περιμένουν να ακούσουν κάτι για τους δικούς και που η Τουρκία με όλους τους τρόπους πραγματικά περιφρονεί, δεν ανοίγει τα αρχεία, δεν επιτρέπει να δοθούν πληροφορίες από τα δικά της αρχεία, παρά μόνο όταν την περασμένη εβδομάδα είχε, ήθελε να γιορτάσει την, σε εισαγωγικά ανακήρυξη του ψευδοκράτους, είχε κυκλοφορήσει ε, βίντεο με τέτοιων υλικών και που έδειχνε, όσοι είχαν την ευκαιρία να το δουν, εχμαλώτους με δεμένα τα μάτια να κατεβαίνουν από λεωφορεία. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι αχμάλωτοι δεν θα περιλαμβάνονται ε, στους αγνοούμενους γιατί θα φρόντισαν να δείξουν μόνο ε, κάποιους που σήμερα βρίσκονται στη ζωή για να μην ε, αυτό από μόνη της παρουσιάσει αγνοούμενους τους οποίους κρατούσε. Όμως είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που έρχονται συνεχώς, όπως την περίπτωση που ανέφερα προηγουμένως την εκταφή οστών από, μαζικούς, από ομαδικούς τάφους, και που η πληροφορία έλεγε ότι δολοφονήθηκε το 1996 ο τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Κουτλού Αταλή ακριβώς για να μην επιτρέψει, να μην ε, του δοθεί η δυνατότητα να διαρρεύσει αυτή την πληροφόρηση στο κοινό. Νομίζω αξίζει τον κόπο να δούμε πώς οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι μαζί μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά που συνέβησαν και το 1974 και δυστυχώς δεν είναι μόνο στρατιώτες που σκοτώθηκαν το 1974 αλλά είναι και άμαχος πληθυσμός και που όπως έχω πει παρουσιάζεται άγνωστη αιτία όπου με εκτελέσεις ε, σκότωναν άμαχων πληθυσμών από παιδιά μέχρι ε, ανθρώπους στα βαθιά γεράματά τους. Γι' αυτό η ευκαιρία που μας έχετε δώσει τούτη είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστούμε και όλα όσα έχουμε να αναφέρει για την ανάγκη στήριξης και της περαιτέρω οικονομικής και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τις χώρες ξεχωριστά και ταυτόχρονα τα δύο άλλα σημεία που ανέφερα, τα αρχεία, τις πληροφορίες, τις στρατιωτικές περιοχές και την επίλυση, αν θέλετε, επιμέρους θεμάτων όπως είναι τα θέματα των πιστοποιητικών θανάτου. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mrs. I think... Σας ευχαριστώ, κύριε του Κουμάκοτρα. Οπωσδήποτε θα έχετε την στήριξή μας και στο μέλλον και όπως είπαμε θα μπει και η πρόταση στην ημερήσια διάταξη των ε, συντονιστών. Λοιπόν, διακόπτουμε τώρα και θα συνεχίσουμε στις 3 η ώρα το απόγευμα. Θα έρθει η Επίτροπος η κυρία Μάλμστρομ που θα παρουσιάσει τρία σημαντικά έγγραφα που ευθύθηκαν σήμερα το πρωί από το Σώμα των Επιτρόπων. Τρεις η ώρα λοιπόν, τα ξαναλέμε. Γεια σας.